σημείο τη σημερινή διάταξης που είναι ο περιορισμός ε, κάποιων ε, ρήπων και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αύριο θα ψηφίσουμε τον ε, ορισμό για πολύ συγκεκριμένους ρήπους και για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και φυσικά τίθενται πολύ συγκεκριμένα όρια. Επίση, Επίσης καλύπτεται ένα κενό νομικό το οποίο το, στη διαδικασία που ορίζει να για τις εγκαταστάσεις ε, καύσης κάτω του 1 ΜΒ και έχουμε και τις εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 50 ΜΒ. Αυτά τα όρια είναι φιλόδοξα γιατί θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα αλλά επίσης ε, θέλουμε να προστατεύσουμε και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τις επενδύσεις ε, κυρίως ε, μέχρι τώρα καλύπτονταν οι μικρές εγκαταστάσεις μέχρι τα 5 ΜΒ. Είναι αυτές οι σημαντικές εγκαταστάσεις ε, για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για τα πανεπιστήμια. Όμως θα πρέπει να καλυφθούν από την νομοθεσία και οι εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας ε, που θα έπρεπε να τροποποιηθούν σημαντικά για να σεβαστούν την νέα νομοθεσία. Επίσης, ε, καλύπτονται και οι εγκαταστάσεις που παράγουν θέρμανση για τα κτίρια Έχουμε ε, εδώ επίσης εγγύηση της παροχής θέρμανσης για τους τελικούς δικαιούχους. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή από περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Ε, πράγματι θέλουμε να προωθήσουμε μια πολιτική αλλαγής, δηλαδή να περάσουμε από την αυτόματη θέρμανση στη συλλογική θέρμανση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Θα ήθελα να σας πω ότι το τελικό κείμενο της οδηγίας αποτελεί μια καλή ισορροπία γιατί αφενός έχουμε την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά από την άλλη λαμβάνουμε υπόψη και την οικονομική πραγματικότητα αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι φιλόδοξοι στόχη αλλά δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε νέο κόστος ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τις επιχειρήσεις. Στις 23 Ιουνίου στον άτυπο τριμερή διάλογο φτάσαμε σε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Εγκρίθηκε και από την Κορεπέρ η συμφωνία αυτή και στις 30 Ιουνίου. Μόνο μία χώρα καταψήφισε και κατόπιν είχαμε την ε, έκθεση στην Επιτροπή, την έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 15 Ιουλίου. 59 ψήφι κατά 6, συγγνώμη, 59 ψήφι υπέρ 6 κατά. Οι διαδικασίες ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες. Αυτή η συμφωνία λοιπόν αποτελεί πραγματικά ένα πακέτο. Το αν αφαιρέσουμε ένα στοιχείο ή αν το τροποποιήσουμε σημαίνει ότι θα έχουμε μία νέα ανάγνωση του όλου σχεδίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, και όλους ε, που με βοήθησαν να διαπραγματευτώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Προεδρία για τη συνεργασία της και για την υποστήριξή της. Ευχαριστώ και την προηγούμενη Προεδρία αλλά και τη σημερινή Προεδρία γιατί κατορθώσαμε να φτάσουμε σε ικανοποιητικέ λύσει για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Φιλ Χόγκεν. Κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικά μέλη του Κοινοβουλίου, με μεγάλη χαρά συμμετέχω εξ ονόματος των συναδέλφων του κυρίου Βέλε, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, σε αυτή τη συζήτηση με σκοπό να μειωθεί η πόλυνση, ιδιαίτερα από μικρές μονάδες καύσης, κάτι το οποίο παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2013. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του προγράμματος ε, του περιβαλλοντολογικού για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα θέμα και ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2013 με την Ιρλανδική Προεδρία. Βεβαίως επιβαρύνει το περιβάλλον, η μόλυνση του αέρα και ήδη ξεκινήσαμε από, τις, ε, ε, από τα συστήματα ανταλλαγή ρήπων. Βεβαίως η σημερινή νομοθεσία συνεχίζει να έχει κενά τα οποία θέλουμε να καλύψουμε. Όπως προτείνεται στην ε, οδηγία για την ανταλλαγή ρήπων υπάρχουν ακόμα και να τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Εδώ ο Επίτροπος Βέλε αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις τροπολογίες που πρότειναν, με την επεξεργασία του κειμένου μπορούμε να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντική πτυχή και ακαιρεότητα αυτού του κειμένου της οδηγίας. Χρειάζεται βεβαίως και κάποια ευελιξία με την πρόταση για τη χρήση βιομάζας σαν καύσιμο και όλες οι προτάσεις ε, οι οποίες συμβαδίζουν με τη βασική μας κατεύθυνση που είναι να διατηρήσουμε υψηλή ποιότητα στον αέρα. Η αποτελεσματικότητα της ε, ενέργειας, οι εκπομπές μονοξυδίου του άνθρακα και οι στόχοι οι οποίοι τίθενται, οι οποίοι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε σε μια βελτιωμένη νομοθεσία να μειώσουμε τα εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να έχουμε συνοχή όσον αφορά τον κύριο στόχο μας που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Πέρα από την περιβαλλοντολογική αποτελεσματικότητα, αυτή η οδηγία προτείνει καινοτομία, νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε στην διαρκώς αυξανόμενη αγορά της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της ρήπανσης. Και βεβαίως σκοπός μας είναι να υιοθετηθεί ταχύτατα και να υλοποιηθεί αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, λέει Πρόεδρος. Και τώρα, εξ ονόματος της Επιτροπής Ήτρε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέντερλη, ο οποίος όμως δεν είναι στην αίθουσα. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν τον ομιλητή εκ μέρους του ΕΛΚ που είναι ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κρυξίπ και όλους τους συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτή της συμφωνίας που μας επιτρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ωρία εκπομπών για ένα τομέα που μέχρι σήμερα δεν είχε ρυθμιστεί. Επίσης ευχαριστώ τον Επίτροπο και την Προεδρία για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής Εξέταση ε, της πρόταση, ε, όπως ε, είπαμε, αφορά τις μεσαίου 150.000 μονάδες με ονομαστική ισχύ από 1 μέχρι 50 ΜΒ, θέτοντα ωριακέ εξίες για τι εφιστάμενε μονάδες καύση και για τις νέες θα μειώσουμε τη ρήπανση και θα έχουμε και ένα σύστημα εγγραφή που θα μας επιτρέπει στα κράτη-μέλη να σεβαστούμε την νομοθεσία. Φυσικά, στόχος είναι να έχουμε την καλή ποιότητα αέρα και να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Το κείμενο αποτελεί ένα συμβιβασμό μεταξύ των διάφορων θέσεων, όμως γενικά πετύχαμε μια συμφωνία που εν μέρη έχει τροποποιήσει την πρόταση της Κομισιόν και βελτίωσε τις δυνατότητες να υλοποιηθεί ρεαλιστικά η οδηγία μέσω της βελτίωσης του ατμοσφαιρικού αέρα ε, Χωρί να έχουμε και υπερβολικό άχθο για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να αξιολογήσουν την δυνατότητα να θέσουν πιο αυστηρά όρια σε ζώνες που δεν σέβονται την ποιότητα αέρα στις Ευρωπαϊκές Ένωση και να υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρηση για να επαληθεύσουμε το 2020 τους προόδου που θα έχουν γίνει ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό ε, ανήκει ε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της COP21 στο Παρίσι. Και εδώ θέλουμε να πούμε ότι φιλοδοξούμε να έχουμε μια συμφωνία φιλόδοξη με την εμπλοκή όλων των μερών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μάσιο Πολούτσι εξ ονόματος των Σοσιαλδημακρών. Επίσης για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τελικά μετά από τόσα λόγια περνάμε και στις πράξεις. Τελικά καλύπτουμε ένα τεράστιο νομοθετικό κενό. Πάνω από 142.000 επιχειρήσεις ε, με ε, τιμές από 1 ως 30 ΜΒ ε, δεν είχαν καλυφθεί. Μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ε, για τη θέρμανση, για την ψήξη, για την παραγωγή ατμού. Μιλάμε για το υδρόθιο, για το ξίδιο του αζότου. Ένα βήμα προς τα μπρος, πολύ σημαντικό για να εντοπίσουμε πιο τελεσματικά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, το υπενθύμησε ο Επίτροπος. Η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη, με από τις κύριες αιτίες ε, ε, ευτροφισμού ε, όπου το βλέπουμε να υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς τα μπρος σίγουρα και μια λογική συμφωνία που υπερασπίζει την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη χωρίς να βλάπτει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εμείς ε, κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές και ας περάσουμε ε, και στην εποπτεία και του μονοξυδίου του άνθρακα. Έχουμε πετύχει μια λογική, ένα λογικό συμβιβασμό ε, για τις ωραίες τιμές και για το χρόνο εφαρμογής. Υπάρχει και υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα για τις ζώνες που δεν σέβονται ε, σήμερα ε, την περιβαλλοντική νομοθεσία και επίσης ε, έχουμε και ειδικές, ειδική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις που παράγουν βιομάζα. Εμείς αύριο θα υπερασπίσουμε ως ομάδα με πεποίθηση αυτή τη νομοθεσία. Σα ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει για την ECR η κυρία Βυσνιεύσκα για δύο λεπτά το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Είναι καλή η είδηση που τελικά διαμορφώνεται με οριστικό τρόπο η οδηγία για τις ε, μεσαίου μεγέθου μονάδε καύση και τι εκπομπέ. Και νομίζω ότι αυτό διασκεδάζει του φόβου που εκφράζονται από διάφορε ε, πηγέ. Οι μονάδε καύση, οι οποίε είναι πολύ ε, δημοφιλείς σε πολλές χώρες όπως και στην Πολωνία όπου βασικά βασίζονται στο κάρβουνο. Αυτό χρησιμοποιείται βασικά στην Πολωνία. Έχουν εξυγχρονιστεί αυτές οι μονάδες στην Πολωνία σύμφωνα με τον νόμο για να υπάρξει περαιτέρω εξυγχρονισμός θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος και αυτό ενδεχομένω να οδηγήσει σε κλείσιμο και να χρειαστούμε τελικά μεμονωμένα συστήματα ε, καύσης που θα οδηγήσει με τη σειρά του αύξηση γιατί μετά δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθούν αυτές οι μονάδες. Και αυτό από πλευρά λοιπόν της ε, υγείας θα ήταν αντιπαραγωγικό. Η δυνατότητα εξαίρεσης ε, τέτοιων ε, μονάδων από τα ανώτατα όρια μέχρι το 2030 αποτελεί μια έκφραση της κοινή λογικής συντελική ανάλυση. Χάρηκα λοιπόν που συμπεριληφθήκε και η δική μου τροπολογία στην τελική μορφή της οδηγίας ότι θα πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις υποσταθερούς όρους όπου και το σκάνδαλο νομίζω της ε, Volkswagen της εταιρείας η οποία εξαπάτησε σε ό,τι αφορά τις εκπομπές σε μια χώρα η οποία είναι τόσο έντονα ταγμένη για την μείωση των εκπομπών, καταδεικνύει ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών. Και επίσης να ελέγχουμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ήδη υπάρχουν. Σας ευχαριστώ από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ο κύριος Χάιτουμα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σκιώδη συγκητή της Άλντε και όλους τους υπόλοιπους σκιώδη συγκητές καθώς και τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες κάψης, ε, μεσαίου μεγέθους, ε, Αυτά η οδηγία έχει ως σκοπό τη μείωση του διοξιδίου θείου, του οξυδίου του αζότου και της σκόνης που έχουν επιβλαβεί σε συνέπειες για την υγεία του κοινού. Με την καλή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε πλέον μια καλή πρόταση στο τραπέζι μας. Εμείς ε, θα θέλαμε οι εξαιρέσει ε, από τα όρια των εκπομπών να μειωθούν στο βαθμό του δυνατού. Αυτό το πετύχαμε και θα πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε ρεαλιστέ, γιατί όταν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την βιομάζα, πρέπει να προσαρμοστεί. Και γι' αυτό έχουν προσαρμοστεί λοιπόν και οι εκπομπέ σε ό,τι αφορά την βιομάζα. επίση ε, να αποφύγουμε τη διπλή νομοθεσία, τη διπλή ρύθμιση. Και αυτό το πετύχαμε. μία εγκατάσταση η οποία έχει ω σκοπό να καλύψει σε περίπτωση κατεπίγουσα ανάγκη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και σε περίπτωση κατεπίγουσα ανάγκη μόνο. Επίση, μειώσαμε την γραφειοκρατία. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφεί κανόνε με ένα ενίο σύστημα διαδότηση. Επίση, είναι καλό το γεγονό ότι θέλουν να μάθουν τα κρατημέλη το ένα από το άλλο. Γιατί σε κάποια κρατημέλη η πρακτική και η εμπειρία είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι σε άλλα. Ε, ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές στην πηγή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα από την GUE NGL η κυρία Μαρτίνε έχει το λόγο. Είμαστε ικανοποιημένοι που πετύχαμε μια συνένεση για την πρόταση αυτή και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ε, εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη και αναφερόμαστε και στις Ασόρες, στα Καναρία, στη Μεδέρα και σε όλη την... στις άλλες ευρωπαϊκές γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το τρίμα κρεφτά αποτελεί εμπόδιο για να αναπνέουν και εκεί οι πολίτες καθαρό αέρα προτιμούμε να προλάβουμε κάποιες εταιρείε να εκμεταλλευτούν νομικά κοινά για να βλάπτουν την υγεία των πολιτών και του πλανήτη. Άλλοι, από ό,τι φαίνεται, θέλουν να υπερσπίσουν περισσότερο τα συμφέροντα των εταιριών παλά των πολιτών που ήταν όταν η Ρεψόλ έκανε τα Κανάρια το κύριο Βενζινάδικο της Ευρώπης. Επίσης, η Κομισιόν ε, πρέπει να ε, αποφυγή να ε, εκπέμπονται κάποιοι ρήποι στην ατμόσφαιρα γιατί είναι ντροπή να συνέβη το αυτό που συνέβη με τη Volkswagen δηλαδή να υπήρχε διποψία ε, για απάτη και να μην έχει γίνει τίποτα μέχρι που ξέσπασε το σκανδαλό ε, το ότι καίγονται ορυκτά καύσιμα αυτό προκαλεί κυρίως τη ρήπανση αλλά ξέρουμε ότι όσοι πλωτίζουν εις ε, βάρος της εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο σε δύο μήνες έχουμε τη Σύνοδο στο Παρίσι και τότε θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ε, θα δούμε τότε ποιος θα πάρει το μέρος ποιου. Ευχαριστώ πολύ. Για ε, τους πράσινους, ο κύριος Σάικου έχει το λόγο. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και καταρχήν εξ ονόματος του που δεν μπόρεσε κυρίας Μίσελ Ριβαζή Θεωρώ ότι ο συγχητής έκανε μια εξαιρετική και πολύ ισορροπημένη δουλειά και εκτούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει το θέμα των εκπομπών. Συζητήσαμε το απόγευμα για την αυτοκινητοβιομηχανία και εδώ μιλάμε για μικρές μονάδες καύσης. Δεν είναι πάντα εύκολο να φτάσει κανείς σε νομοθεσία όταν μιλάμε για ποιότητα του αέρα γιατί οι περισσότεροι λένε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε την αιτία, δηλαδή να καταπολεμήσουμε την πηγή της ρήπανσης. Και βεβαίως εδώ δεν θα πρέπει απλώς να ασχοληθούμε με επέκταση των προθεσμιών, με αναβολές, με τρόπους να παρεκκλίνουμε διότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και σε αυτή την νομοθεσία όπως και σε άλλες. Βλέπω όμως ότι με μεγάλη χαρά αυτή τη φορά το Κοινοβούλιο δεν υποχώρησε και δεν υπέκυψε στις πιέσεις να υπάρξουν αναβολές και εξαιρέσεις. Όσον αφορά τα ανώτατα όρια, τέθηκαν με αποφασιστικότητα. Κάθε φορά όμως που μιλάμε για ποιότητα του αέρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο αποφεύγεται, αλλιώς θα είμαστε πάντα μακριά από το στόχο μας που είναι βελτίωση της ποιότητας του αέρα, που είναι και ο στόχος των καταναλωτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους όσοι συνεργάστηκαν και δεχόμενο το Συμβούλιο που θα μπορούσε να είχε συνεργαστεί περισσότερο. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Έσεριτς. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε τόσο αργά αυτή την μπλε κάρτα. Πολύ σύντομα. Μιλήσατε για πηγή, για αιτία της ρήπανσης. Εδώ όμως βεβαίως μιλάτε για την βιομηχανία. Χωρίς τη βιομηχανία δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθούν οι φιλοδοξίες σας για καλύτερο ποιοτικά αέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί προς τη βιομηχανία, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης. Εύκολη είναι η ερώτησή σας. Αν με ακούσατε, θα διαπιστώνατε ότι ήμασταν πολύ φιλικοί προς τη βιομηχανία. Διότι σήμερα πληρώνουμε δισεκατομμύρια για να θεραπεύσουμε τις ασθένειες που προκαλεί η ρήπανση του αέρα. Αυτή όμως που τελικά μολύνουν, ρηπαίνουν, θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θεραπεύουν και χρηματοδοτούν και όχι όλοι εμείς η κοινωνία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πετιτσίνη έχει το λόγο για ένα, λεπτό, για ένα λεπτό. Είναι αλήθεια ότι με την πρόταση αυτή καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό για τη για τις μονάδε καύσης που δεν ε, είχαν καλυφθεί μέχρι τώρα με την νομοθεσία Όμω δεν μπορούμε να εκδεστήσουμε το κενό με το τίποτα. Εδώ δεν υπήρχε καμία βούληση να βάλουμε ιδιαίτερα τοξικού ρήπου όπω το, οι διοξίνε. Έτσι λοιπόν ε, είναι ελλειπή αυτή η οδηγία. επίση. έχει αποδυναμωθεί η πρόταση τη Κομισιόν λόγω τη παρέμβαση του Κοινοβουλίου αλλά έχουν αποκλειστεί και οι offshore πετρελαϊκές πλατφόρμες και οι εγκαταστάσεις που κάνουν βιομάζα και μπορεί να ρηπαίνουν χωρίς όρια. Και αν μιλάμε για την πραγματική ανταγωνιστικότητα, ε, ε, πρέπει να δούμε και την δυνατότητα οικολογικής καινοτομίας, δηλαδή να χρησιμοποιούν τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα για μια ακόμη φορά εξυπηρετούμε τις πετρελαϊκές πολυεθνικές και τη βιομηχανία που παράγει ηλεκτρισμό. Σας ευχαριστώ που με εγκεκριμένους. Ο κύριος Μπάλτσο για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όταν συναντηθήκαμε τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει σε διεθνή φόρα τη δέσμευσή της για τη μείωση των ρηπαντών που εκλείονται στην αέρα μας, στην ατμόσφαιρά μας και θέλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα στις τρίτες χώρε. Θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι στη δήλωση, για τη δήλωση αυτή. Αλλά ας δούμε τι έγινε με τη Volkswagen. Ωραία τα λόγια, αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει έκπληκτοι από αυτό που συνέβη με την Volkswagen. Ποιε είναι λοιπόν οι υποχρεώσει μα, Οι υποχρεώσει μα δεν ε, είναι να προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα. Είναι σημαντικό αυτό να μπει στην οδηγία και είναι σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον ε, στοιχείο για τη ρήπανση της ατμόσφαιρας στο γεγονός ότι τόσοι πολλοί πολίτες της Ένωσης επηρεάζονται από τη ρήπανση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχάρει τον εισηγητή και χαίρομαι που υπάρχουν τροπολογίε αυτέ ε, και χαίρομαι που τι υποστηρίζει και ο εισηγητή δεν θα μπορούσε να υποστηρίξω το κείμενο χωρίς αυτέ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχαϊρπιερικ, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Επίτροπε, ευχαριστώ τον εισηγητή και για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει σε αυτό το τεχνικό ζήτημα, το οποίο ωστόσο είναι εξίσου πολιτικό. Σήμερα μιλάμε για τη μείωση των εκπομπών κάποιων ε, ε, ρηπαντών από μεσαίου μεγέθους μονάδες κάψης ε, στις Ήπετρο στις πόλεις σε μονάδες που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Στην Ευρώπη έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο για την, ε, για την ε, βελτίωση της ποιότητας ε, της ατμόσφαιρας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει καλή νομοθεσία, καλή νομοθεσία για την δημόσια υγεία, για την ρήπανση. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήνουμε ανοιχτή την πίσω πόρτα για να φροντίσουμε τα συμφέροντα κάποιων. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να κοιτάξει κατά πόσο πρέπει να αλλάξουν οι οριακές τιμές βάσει των καινούριων τεχνολογιών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βέλτιστες, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν όρια παρόμοια με αυτά του παρελθόντος αν ε, βελτιωθεί η τεχνολογία στο μέλλον. Γιατί η καινοτομία κινείται γρήγορα, αλλά πολλές φορές δεν κινείται εξίσου γρήγορα η φιλοδοξία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την εφαρμόσιμότητα και τις οικονομικές συνέπειες και την απασχολησιμότητα σε ό,τι αφορά τη μεγάλη κλίμακα οικονομικών επιχειρήσεων θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη δεν θα πρέπει να είμαστε λοιπόν τυφλοί και φανατισμένοι για να μην κάνουμε διακρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν πολλές ε, ομάδες ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τάχθηκαν υπέρ κάποιων εξαιρέσεων σε κάποιες περιπτώσεις όπου η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι ήδη αρκετά καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πολύ. Ο κύριος Παρνιό έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την ΚΑΠ 21 στο Παρίσι και πραγματικά η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι στην καρδιά αυτών που θέλουμε να προωθήσουμε. Η βελτίωση του αέρα που αναπνέουμε δεν μπορεί παρά να είναι ένα σημαντικό στόχος. 348.000 θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε κακή ποιότητα του αέρα. Κινδυνεύει η υγεία μας από αυτή τη μόλυνση και γι' αυτό και ιδιαίτερα συγχαίρω τον εισηγητή γιατί πετύχαμε πολύ σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά ρήπους, το διοξίδιο του αζότου, το μονοξίδιο του άνθρακα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό σε άλλα νομοθετικά κείμενα. Και αυτό ζητούμε από την Επιτροπή. Εν ώψη λοιπόν της ΚΑΠ 21 πιστεύω ότι η έκθεση αυτή μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα τρόπο καταπολέμησης της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζούλη Γκόλινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Εκ μέρου τη αντιπροσωπεία μου θέλω, τη ομάδα μου, θέλω να καλωσορίσω αυτή τη συμφωνία. Ξέρω ότι ήταν δύσκολε οι διαπραγματεύσει και εδώ έχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ αποκλίνουσων απόψεων και θέλω να δράξω την ευκαιρία για να συγχαρώ ιδίω τον εισηγητή για τις δεξιότητες του. Εμεί ε, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε μια συμφωνία και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο. Η κακή ποιότητα του ΜΕΡΕ είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ζητάμε για την τελειότητα, όμω η τελειότητα, το τέλειο είναι το, ο εχθρό του καλού. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα εδώ να δούμε και και το ρεαλισμό και να έχουμε συνθήκε που θα μα επιτρέψουν να έχουμε επενδύσει, νέε τεχνολογίε νέες ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Στόρβαλτς. Για ένα λεπτό έχει το λόγο τώρα. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητάμε τα θέματα τη ε, ποιότητα τη ατμόσφαιρα ε, όλη την ημέρα σχεδόν από διαφορετικές οπτικές ε, γωνίες. Αυτό καταδεικνύει την ανησυχία και την εύλογη ανησυχία μας. Πρωτού φύγω για το Στρασβούργο, είδα ένα ενδιαφέρον μας στη Φιλανδία από τη Λαπωνία συγκεκριμένα, που είναι η πιο καθαρή περιοχή σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Όπου είναι δύο άτομα ανά χιλιόμετρο η πυκνότητα του πληθυσμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ισορροπημένος ο συμβιβασμός που ε, επιτεύχθηκε για να πετύχουμε την ε, μείωση των εκπομπών, αλλά θα πρέπει να μην ε, ακολουθήσουμε τη μία λύση για όλους απαραίτητα. Η Λαπωνία αποτελεί ένα καρό παράδειγμα. Πιο πολλοί θα ξέρουν ότι έχουμε κρύους χειμώνες στη Λαπωνία. Είναι και ο Άι Βασίλης, ξέρετε, με το ελκυθρό του που έρχεται. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό σα βράδυ. Σα ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Δεν έχουν ακόμα φτάσει τα Χριστούγεννα, ωστόσο. Επόμενη ομιλητρία, η κυρία Κονέτσνα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και τα Εθνικά Κοινοβούλια, έχουν ε, ασχοληθεί με τα όρια εκπομπών ορισμένων ε, εγκαταστάσεων ε, για πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα Έχουμε καλύψει και τις μονάδες κάτω των 50 ΜΒ, όμως πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, όπως για το όριο του υδρόθεου. Πήγαμε πολύ μακριά γιατί σε ορισμένες χώρες μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Παίρνουν τους χάρη να το να κλείσουν μικρές εγκαταστάσεις ε, παραγωγής ε, θερμότητας ε, μπορεί να οδηγήσει στην μεγαλύτερη χρήση λιγνίτη. Ελπίζω λοιπόν ε, ότι θα πρέπει να δούμε και ε, τις τοπικές εγκαταστάσεις ε, και δεν αναφέρουμε μόνο στις μονάδες στην Τσεχία αλλά και στις συνοριακές περιοχές, τους χάρη και στην Πολωνία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε δίκαιοι προς αυτή την κατέντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα κυρία Τζούλια Ρίνη για ένα λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, η ομάδα μου πιστεύει στην σημασία της ε, βελτίωσης της ε, ποιότητας του αέρα, αλλά είμαστε κατά της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Είμαστε αντίθεση με την οδηγία για την οικολογικό σχεδιασμό και για την οδηγία ε, για τη μείωση των εκπομπών και θα είμαστε λοιπόν κατηγορηματικά κατά και της οδηγίας αυτής για το μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται σε ό,τι αφορά επίση την καταχώρηση των νέων εγκαταστάσεων. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επαφείται στους ευρωκράτες των Βρυξελών. Και θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει υπερβολική ρύθμιση, γιατί οι τρέχουσες νομοθεσίες δεν έχουν δώσει νομική βεβαιότητα στους επενδυτές. Η υπερβολική ρύθμιση απειλεί τις επενδύσεις στην παραγωγή, την ελευθερία αγορά και η επιπρόσθετη ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν πρόκειται να προωθήσει την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Θα πρέπει να είναι αγωνιστική και να αυξήσει την παραγωγικότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρη για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε πίτροπε, η ρήπανση στον αέρα σαφώς και επηρεάζει τη γενικότερη ρήπανση του περιβάλλοντος αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Στα πλαίσια των προσπαθειών να μειωθούν οι πρόοροι θάνατοι, οι οποίοι έφτασαν τις 400.000 το 2010, το σύνολο των δαπανών ξεπερνούν το ποσό το οποίο είχαμε αρχικά προβλέψει. Και εδώ αναφερόμαστε και σε ποσά για την... Ε, για τον τομέα των κατασκευών, για την ανανέωση κτίριων που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Βλέπουμε σήμερα ότι τα προβλήματα της μόλυνσης του αέρα είναι πάρα πολύ οξία στην Ευρώπη. Επί δεκαετίες εργάστηκα στον τομέα αυτό στη χώρα μου για μικρό, μικρούς ε, και μεσαίες μονάδες καύσης και τη ρύθμιση αυτών και διαπιστώνουμε ότι εδώ στη Βοσνία Ζεγοβίνη υπάρχει σημαντική ρήπανση η οποία οφείλεται στις γειτονικές χώρες. Έχουμε λοιπόν σοβαρά προβλήματα από ρήπανση την οποία δεν προκαλούμε εμείς αλλά οι γειτονικέ μας χώρες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές και πρότυπα για τις ε, μικρομασίες αυτές μονάδες καύσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρλος Ορίνιο για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Πίτροπε, Έχουμε πάρα πολύ σημαντική νομοθεσία και λόγω της επόμενης συνόδου κορφής ε, για το κλίμα, ε, Καλώς ε, έχουμε και την πρόσφατη κρίση με τα οχήματα. Θα πρέπει να έχουμε ε, ηγετική θέση για να προστατεύουμε την ποιότητα του αέρα και θα πρέπει η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της στην βιώσιμη και πράσινη οικονομία. Το να έχουμε ποιότητα του αέρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα. Πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για ε, μια τεχνολογική ηγεσία. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα θέματα και πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και για μας αλλά και απέναντι στον κόσμο. Θέλω να τονίσω και τα χαρακτηριστικά αυτής της οδηγία σε ό,τι αφορά τη απλούστευση τη διαδικασία, γραφή, και χορήγηση αδειών. Σας ευχαριστώ. Ο για ένα λεπτό είναι Πρόεδρε, Επίτροπε, όπως ε, καταδεικνύουν και οι μετρήσεις σε κάποια κρατημέλη, σε κάποιες χώρες ε, υπάρχει μεγάλη ρήπανση της ατμόσφαιρας και αυτό φυσικά επηρεάζει και τις ε, ε, περιοχές, τις περιοχές μάλλον που είναι κοντά στα σύνορα και αυτό ασφαλώς λοιπόν επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα της ατμόσφαιρας και σε γειτονικέ χώρες. Είναι δύσκολο να μετρηθούν οι μικρές μονάδες καύσης. Ωστόσο, τα όρια που θα πρέπει να επιβληθούν και στις μικρές αυτές εγκαταστάσεις είναι σημαντικά αν θέλουμε να περιορίσουμε τις ρήπαντες. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει μια συνεχτική προσέγγιση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο οι κανόνες που επιβάλλονται, αλλά και πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονιστούν αυτές οι μονάδες, είτε υποστηρίζοντας την καινοτομία ή υποστηρίζοντας και την έρευνα πιο σύγχρονων μέσων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόταση αυτή. Κάτι όμως πραγματικά δεν κατανοώ. Γιατί αποκλείονται οι περιφερειακές περιοχές οι πολύ στις περιοχές. Σίγουρα κάποια ομάδα πίεσης ε, θα οδήγησε σε αυτόν τον αποκλεισμό, τον οποίο εμείς βεβαίως απορρίπτουμε, καθότι οι απομακρυσμένες αυτές περιοχές και παραμεθόρεις θα αποκλειστούν και δεν θα ισχύουν για αυτές τις ε, παραμεθόριες, για αυτές τις νησιωτικές και άλλες περιοχές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα, αυτές τις περιοχές και το άρθρο 341 σήμερα χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε. Έχουμε υποβάλει λοιπόν ξεχωριστές τροπολογίες και καλό όλους να τις υποστηρίξουν αύριο. Ο κύριος Έσερτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε μία νέα οδηγία για να καταπολεμήσουμε την ε, ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας ε, στα Μίτλαντς. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται η Μαύρη Χώρα και εκεί ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν μαύρος ο αέρας με νέφος και πάρα πολλοί άνθρωποι στην περιοχή μου πέθαναν από τη ρήπανση. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνω την απέτηση για καθαρό αέρα. Βέβαια με το πέρασμα των χρόνων δεν ισχύει κάτι γιατί η αποβιομηχανοποίηση ε, αλλά και τα μέτρα τη κυβέρνηση οδήγησαν στον καθαρισμό του αέρα. Δεν πιστεύω ότι ο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να υποκείμεθα σε έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι από μόνοι μας μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό, αλλά πιστεύω ότι όποιο και να το διαχειριστεί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό να μην ε, πάρουν μέτρα που να ε, καταστήσουν πιο δύσκολη την κατάσταση για τη βιομηχανία. Δεν ε, πρέπει να αυτοτιμωρούνται πλέον οι οικονομίες μας. Έτσι λοιπόν, προσοχή, αυτό θέλω να τονίσω και το ΕΒ μπορεί να τα καταφέρει και μόνο του. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Λουκασιεύσκα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σίγουρα η πολιτική μας στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, καθοριστικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της κρίσης, έχει σήμερα σημαντική εμβέλεια και είναι βεβαίως και μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι η εκπομπή ρήπων ουσιαστικά οδηγεί σε περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους. Βλέπουμε ότι η εκπομπή αυτών των ρήπων ουσιαστικά φτάνει μέχρι και 900, 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βλέπουμε ότι εδώ χρειάζεται μια μεγάλη διαβούλευση και υποβολή προτάσεων Αναρωτιέμαι αν σήμερα δεν επιβάλλουμε πάρα πολύ αυστηρούς στόχους. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τι έγινε με την επιβολή στόχων που δεν εφαρμόστηκαν και την υπόθεση Volkswagen. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον εισηγητή γιατί πραγματικά έλαβε υπόψη του όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όλους τους φορείς. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας, αλλά και για όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη λογικοί στόχοι, με προσοχή και βεβαίως ε, και η σκόνη αλλά και το διοξίδιο του άνθρακα που σαφώς πλήττουν και το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία να ληφθούν υπόψη και να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι και την ίδια ώρα να αποφευχθεί περιττό γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως να μειωθεί και το κόστος για τον τελευταίο καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάντεν, το λόγο για ένα λεπτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για αυτή τη συζήτηση η οποία σήμερα είναι κατανοητή κατά την άποψή μου για τους Ευρωπαίους. Ποιοι είναι οι στόχοι, τι θέλουμε να πετύχουμε. Πρόκειται εδώ για πιο καθαρό αέρα και να αποφύγουμε 400.000 άτομα το χρόνο να χάνουν τη ζωή τους λόγω ασθενειών που προκαλούνται από ασθένειες που οφείλονται σε αυτή τη μόλυνση, καρκίνους κυρίως. Μεταξύ 330 και 900 εκατομμυρίων ευρώ είναι το κόστος που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν είχαμε καλύτερη πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος. Βεβαίως δεν μπορούμε διαμιάς να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά οι στόχοι που τίθενται είναι στόχοι που οφείλονται και είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, ρεαλιστικών συμβιβασμών, από τη μία λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και την υγεία των Ευρωπαίων και από την άλλη τις ε, απαιτήσει της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Μπογκανίεβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του κ. Τζίπα αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. θέμα την έλλειψη ε, νομοθεσίας για τις ε, μόνατε κάψει μεσαίου μεγέθου που προκαλεί παραθυράκια στην νομοθεσία μας και προβλήματα από πλευρά ε, του νομοθέτη. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τις εκπομπές ρηπαντών στην ατμόσφαιρα, αλλά η υπερβολική ρύθμιση καταστά δύσκολη την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και επίσης συνδέεται με πολύ πρόσθετο κόστος. Εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηρή νομοθεσία, ενώ άλλοι ρηπαντές όπως η ΙΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία κοφεύουν σε ό,τι αφορά τις προτάσεις ε, εφαρμογής παρόμοιων προτύπων στις χώρες τους. Αυτό φυσικά καθιστά δύσκολη τη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και μειώνει και τις ε, θέσεις απασχόλησης. Να προσέχουμε λοιπόν όταν συζητάμε τέτοιες ε, προτάσεις, προκειμένου να μην υπάρχει αναποτελεσματικότητα και επιπρόσθετο κόστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπόιλαν, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά το γεγονό ότι διαφωνώ με τον αριθμό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην έκθεση, καλωσορίζω την νομοθεσία εν για την ε, εκπομπή λοιπόν από μεσαίου μέγεθους μονάδες καύσης. Γίνεται λοιπόν ε, πληρώνεται αυτό το χάσμα επιτέλους μεταξύ μεγάλων και μικρών μονάδων ε, καύσης. Στην Ιρλανδία 1300 θάνατοι ε, σχετίζονται με την φτωχή ποιότητα της ατμόσφαιρας. 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αυτό κοστίζει φυσικά και στον πολίτη την υγεία του και στην, ε, στον εθνικό προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίζουμε να κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα όρια ε, του διοξιδίου του θείου και τα οξύδια του αζότου στην Ιρλανδία, μας καταδεικνύουν πόσο κατεπίγουσα είναι η ανάληψη δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για δύο λεπτά για το λόγο κύριο Σόγκαρο. Ευχαριστώ πολύ. Παρά την μεγάλη πρόοδο που γίνεται για την αντιμετώπιση της ρήπανσης ε, της ατμόσφαιρης σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου θείου, του και σκόνης, ε, υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά αυτά που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και έτσι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και για την υγεία μας. Και αυτό έχει ασφαλώς αντίκτυπο και ε, στο, στα οικονομικά μας. Εκατοντάδες ε, δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει η εκπομπή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που καλύπτεται αυτό το κενό μεταξύ μικρών και μεγάλων μονάδων καύση και αποφεύγουμε την αλληλεπικάλυψη στην νομοθεσία. Περίπου 7% από τις ε, μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης είναι στα χέρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι σημαντικό να μην επιβαρυνθούν υπερβολικά και αυτές οι επιχειρήσεις. Και πιστεύω λοιπόν ότι η ισορροπία που βρέθηκε είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ του εφικτού και του περιβαλλοντικά ευλογού σε ό,τι αφορά τα συστήματα θερμάνσης ε, εξαπόστασης και άλλα συστήματα. Είμαι επίση ικανοποιημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία πει για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για να το συζητάμε τόσο αργά τη νύχτα. Δυστυχώ τα τελευταία δέκα χρόνια δεν βελτιώθηκε η κατάσταση και κάθε χρόνο οι θάνατοι είναι πάρα πολύ και τα αναπνευστικά προβλήματα στις πόλεις είναι πολύ μολυσμένος ε, ο αέρας και φυσικά εδώ μιλάμε για ένα συμβασμό. Πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα μέχρι και που είναι δυνατόν. Στην Ευρώπη είναι αλήθεια ότι η ποιότητα του αέρα είναι χειρότερη σε ορισμένε περιοχέ από άλλε. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ε, δηλαδή να έχουμε ριζικά μέτρα για τη βελτίωση της ε, ποιότητα του αέρα. Φυσικά όμως εδώ βλέπουμε να έχουμε μεγάλε μεταβατικέ ε, περιόδους για όσου ε, έχουν ε, προβλήματα για τι επιχειρήσει που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Νομίζω ότι τελικά έχουμε μια ισορροπημένη λύση και μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους όσο το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε όλα αυτά ε, σεβόμενοι και τις ε, βιομηχανίες. Ε, Ο Κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή την νομοθεσία που είναι πάρα πολύ σημαντική καλύπτεται ένα νομικό κενό σε σχέση με τις μεσές μονάδες καύσης από ένα ως 50 ΜΒ που δεν είχαν ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν το 80% του συνόλου και χρησιμοποιούνται για πάρα πολλές εφαρμογές και παράγουν σχεδόν το 1 τρίτο των εκπομπών υδρόθιου, των οξυδίων του αζότου και σωματιδίων. Η ρήπανση του αέρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών και στο κόστος των εθνικών συστημάτων υγείας. Στο τελικό κείμενο και χάρη στην δουλειά που έγινε από τον συγητή, που τον ευχαριστώ, αλλά και χάρη στο σκιώδη συγητή μας, τον Μάσιμο Πολούτσι και τον Υπουργό εγκαλέται κατά την Τελική Προεδρία ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε μία φιλόδοξη πρόταση που αν εφαρμοστεί και στις εφιστάμενες αλλά και στις νέες μονάδες θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης χωρίς παρόλα αυτά να θέσει υπερβολικά αχθή στις επιχειρήσεις μας. Und nun ist im Rahmen des ο κύριος ε, Ρικάρδο Σάντος στη διαδικασία Κατσβιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτή η νομοθεσία είναι ευπρόσδεκτη και μας δείχνει τις προσπάθειες να υπάρχουν συνέργειες ε, για την ποιότητα του αέρα, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη μετριασμού των παγκοσμίων κλιματικών αλλαγών. Οι προτάσεις ε, θα υποχρεώσουν ε, να έχουμε όρια εκπομπών που προτείνονται από την Κομισιόν Επίσης είναι θεμελιώδες ε, η εξαίρεση των υπερπόντιων εδαφών εδώ. Αναγνωρίζουμε ε, τον ισιωτικό χαρακτήρα ε, και ίσως ότι πρέπει να δοθούν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτές τις περιοχές. Οι Ασόρες, από όπου προέρχομαι εγώ, αποτελούν ένα παράδειγμα πάρα πολύ θετικό σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, χάρη σε, μια συνεχή δέσμευση της φυσικής κληρονομιάς. Αυτή είναι μια διαδρομή που θα συνεχίσουμε να την διατρέχουμε με περηφάνεια. Σας ευχαριστώ. Της Μάριας, Ο συνάδελφοι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ενημερώσω για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους δύο χειμώνες η πατρίδα μου η ελλάδα λόγω της εθαλομύχλης που έχει εμφανιστεί στις ελληνικές πόλεις και ειδικά στην αθήνα και τη θεσσαλονίκη. η εμφάνιση της εθαλομύχλης οφείλεται αποκλειστικά στο μνημόνιο που επέβαλε την αύξηση των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος και οδήγησε έτσι χιλιάδες συμπολίτες μου στην αναζήτηση μεθόδων θέρμανσης του προπροηγούμενου αιώνα όπως αυτοσχέδια μαγκάλια και καύση κάθε είδους ακατάλληλης καύσιμης ύλης. η μέθοδοι αυτή είναι άκρως επικίνδυνη για τους ίδιους τους πολίτες και για τη δημόσια υγεία. για τους λόγους αυτούς καλώ την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει άμεσα την επιβολή μηδενικού ΦΠΑ και να μειώσει στο ελάχιστο τον φόρο κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης διαφορετικά ο ελληνικό λαός θα παγώσει και αυτό το χειμώνα και θα βρεθούμε και φέτο αντιμέτωποι με την υγειονομική βόμβα της εθαλομύχλη με ευθύνη αποκλειστικά της τρόικα και της συγκυβέρνησης σύριζα ανέλ. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. για ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω αυτήν την έκθεση καθότι περιορίζει τις εκπομπές και είναι πολύ σωστό βεβαίως να υπάρχουν εξαιρέσεις για μετά το 2030 για μονάδες κάψεις που λειτουργούν με βιομάζα. Για γεωπολιτικούς λόγους χρειάζεται μετάβαση μέχρι να υιοθετηθούν πλήρως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι μονάδες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμα συμβατικά καύσιμα θα πρέπει να έχουν κάποια ευελιξία και ζητώ από την Επιτροπή να δώσει κάποιο χρόνο σε αυτές τις μονάδες έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβιβαστούν και να συμμορφωθούν με τα νέα πρότυπα. Χρειάζεται μία μετάβαση και μην ξεχνάτε ότι όλος αυτός ο τομέας δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ανεξαρτησία στην ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πολλοί από εσά υπογράμμισαν την οδηγία για τις μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους που θα βελτιώσουν σαφώς ε, την πολιτική μας ε, στον τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Μιλήσατε για την βιομάζα και για άλλες μεθόδους που βεβαίως δεν είναι σε καμία περίπτωση οι ιδανικές. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε το κείμενο, δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να βελτιωθεί και να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες μονάδες καύσης. Δίνονται κάποια περιθώρια για τη χρήση βιομάζας και σκοπός μας είναι σήμερα να δούμε πώς η οδηγία αυτή θα μπορέσει να εφαρμοστεί στις μεσαίες μονάδες καύσης. Νομίζω ότι και ο εισηγητής και όλοι όσοι έχουν συνεισφέρει στο κείμενο αυτό προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένας από τους στόχους αυτού του κειμένου. Κοιτούμε λοιπόν ποια είναι τα συνοδευτικά μέτρα για να μπορέσει να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνονται προθεσμίες και βεβαίως μειώνονται ε, οι απαιτήσει ε, για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις μικρές μονάδες καύσης. Βλέπουμε ότι βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες κάποιων περιοχών. Και το προτείνει αυτό η Επιτροπή στις ε, περιοχές της. Λαμβάνουμε υπόψη επίσης και τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και σε αυτές τις περιοχές υιοθετώντα κριτήρια τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο στην ε, υπηρετική Ευρώπη και στα πολύ απομακρυσμένα νησιά. Είναι αυτό κάτι που πρέπει να το προσαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους έχουν συνεργαστεί με τον εισηγητή και βεβαίως εξ ονόματος του Επιτρόπου Βέλε θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί θεωρώ ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη είναι εξαιρετικά σημαντικός και γενικός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω στο εισηγητή το λόγο. Ναι, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Ακριβώς για αυτό που μόλις είπε τώρα. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που οφείλεται στη δουλειά όλη τη διαπραγματευτική ομάδα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικού περιβαλλοντικούς στόχους που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα και θα συμβάλλουν και στη μείωση των νόσων που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Πρόκειται για ένα συμβιβασμό που λαμβάνει υπόψη και τα οικονομικά συμφέροντα των διάφορων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά επίση ε, προστατεύονται και τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών που ίσως να έχουν προβλήματα για τη διατήρηση αυτών των μονάδων καύση. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Λαβία που καθόλου τη διαπραγματευτική διαδικασία στον τριμερή διάλογο ήταν παρόν, συμμετείχε και υπενθύμησε ότι και τα κράτη-μέλη μπορούν να εισαγάγουν πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με το τι προβλέπει η οδηγία βάσει καλύτερων τεχνολογιών που μπορεί να έχουν στη διάθεσή του. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη δεν είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ε, τη δική τους πολιτική. Μπορούν να το κάνουν, μπορούν να προχωρήσουν κατά αυτόν τον τρόπο και μπορούν να παρέμβουν όταν αυτό χρειαστεί απαραίτητο στις περιπτώσεις που η ατμοσφαιρική ρήπανση υπερβαίνει κάποια όρια. Η εισαγωγή κάποιων παρακλήσεων, κάποιων εξαιρέσεων είναι λογική. Έχουμε λάβει υπόψη την δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων, παραδείγματος χάρη εκεί που είχαμε να κάνουμε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκεί που χρησιμοποιεί τη βιομάζα. Η βιομάζα παράγει περισσότερη σκόνη. Επομένως, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα να θα έχουμε νέες εγκαταστάσεις ή μηχανισμούς για να μειώσουμε την παραγωγή αυτής της σκόνης. Τότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε την φυστάμενη μονάδα καύσης μέχρι τον τεχνικό του θάνατο, εάν θέλετε, έχοντας κατά νου στη συνέχεια στο μέλλον να οικοδομηθούν νέες μονάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο και τους ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν για την επίτευξη αυτού του ισορροπημένου αποτελέσματος. Και ευχαριστώ και όλους που υποστήριξαν τις προσπαθίες μας. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά και ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό.